Jó kívánok, hölgyeim és uraim! Κυρίε και κύριοι, αξιότιμοι ευρωβουλευτέ, κύριε Επίτροπε, μετά από μια πολύ σύντομη διακοπή, συνεχίζουμε τις εργασίες της Συνόδου. Το πρώτο σημείο της ημερήσιας διάταξης για το βράδυ είναι μια δήλωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κατάσταση στην Αλβανία. Θα ήθελα εν είδης να δώσω το λόγο στον Επίτροπο Στέφαν Φίλε για να μας κάνει τη δήλωση της Επιτροπής. Uh, uh, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη. Thank you for inviting me to speak. Uh, σας ευχαριστώ που με καλέσατε να σας μιλήσω για την Αλβανία απόψε. Παρόλο που ήταν απομονωμένη στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο για το μεγαλύτερο διάστημα του 20ου αιώνα η χώρα, σήμερα είναι ανοιχτή και προσιτή. Είναι πλέον μια χώρα με ευρωπαϊκή προοπτική. Σήμερα η Αλβανία βρίσκεται σε μια πολιτική κρίση. Τα γεγονότα στα Τύρανα την Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2011 ε, ήταν πολύ τραγικά. κλιμακώθηκε η πολιτική όξυνση και οδήγησε σε τέσσερις άσκοπους θανάτους. Πρέπει να αλλάξει το ύφος και ο τόνος ε, της αντιπαράθεσης στα τύρανα. Θα πρέπει να σταματήσει αυτή η κλιμάκωση της βίας και να λυθεί η πολιτική κρίση. Αυτό είναι κοινή ευθύνη όλων των πολιτικών ηγετών της Αλβανίας. Αυτό άλλωστε είναι και εκείνο που αναμένουν οι πολίτες της Αλβανίας. Και έχουν δίκιο. Οι δημοκρατικά εκλεγμένοι εκπρόσωποι θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες και το ρόλο τους. Να εκπροσωπούν το λαό και να βρίσκουν δημοκρατικούς συμβιβασμούς. Πρόεδρε, η λύση του προβλήματος θα δοθεί από τους Αλβανούς τους ίδιους. Εμείς ως εξωτερικοί το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να διευκολύνουμε την εξέβρεση μιας τέτοιας λύσης. Η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ε, και ο αντίστοιχο ε, διευθυντή Φλάιτσεκ δύο φορέ επισκέφθηκε τα Τύρανα για να συναντηθεί με τον πρόεδρο, τον πρωθυπουργό και τον ηγέτη τη αντιπολίτευση. Και ε, χαίρομαι που σήμερα ε, είναι μαζί μου το μήνυμα της ΥΠΑ, εκπροσώπου και αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της κάθε, άστον, της και μου είναι σαφέστατο. Πρώτον, να σταματήσει η βία και να διερευνηθούν τα γεγονότα ε, της 21ης Ιανουαρίου με σωστό τρόπο. Οι έρευνες αυτές θα πρέπει να γίνουν από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές χωρίς πολιτική ανάμειξη. Δεύτερον, να σταματήσουν ή ε, φραστικές ε, αντεγκλήσεις ε, ρητές και υπενιγμοί που υπονομεύουν τους πολιτικούς θεσμούς. Τρίτον, θα πρέπει να επανέλθει ο πολιτικός διάλογος. Να αναγνωρίσουν ότι έχουν κοινή ευθύνη για να εγγυηθούν ένα πιο θετικό μέλλον στην Αλβανία. Στο εγγύς μέλλον αυτό σημαίνει από κοινού διασφάλιση ε, της δεξαγωγής ελευθέρων ε, σωστών και διαφανών τοπικών εκλογών. Στη συνέχεια, θα πρέπει να αρχίσει η σημαντική άσκηση εφαρμογής των 12 προτεραιοτήτων, όπως αυτές ορίζονται στη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2010. Η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση είναι υποχρεωμένες να συνεργαστούν στην προσπάθεια αυτή. Οι πολιτικοί ηγέτες και ε, ε, ο λαός έδωσαν θετικά μηνύματα στο διευθυντή που επισκέφτηκε τη χώρα. Τώρα υπάρχει μια ευκαιρία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και που πρέπει να αξιοποιηθεί έτσι ώστε η κρίση να γίνει ευκαιρία. Οι δύο Αλβανοί ηγέτες καλωσορίζουν την προσοχή που τους δίδουμε, αλλά βρίσκονται εγκλωβισμένοι στο εσωτερικό τους αδίέξοδο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει και καλή βούληση, έχει και ε, βοήθεια που παρέχει, αλλά αυτό δεν μπορεί να αντικαταστήσει ούτε να υποκαταστήσει το διάλογο μεταξύ των ηγετών. Εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε να γεφυρωθεί το χάσμα με ενεργή ε, συμμετοχή. Ωστόσο, δεν μπορούμε να το πράξουμε πριν δείξουν αυθεντική και γνήσια βούληση οι δύο πλευρές να βάλουν ε, το ευρωπαϊκό μέλλον της Αλβανίας πάνω από κομματικές σκοπιμότητες και προσωπική καχυποψία. Δεν υπάρχει χώρος τώρα για χρονοτριβές. Θα πρέπει η Αλβανία να ανταποκριθεί σε όλα τα κριτήρια της Κοπενχάγης και μεταξύ αυτών είναι ο διαδραστικός πολιτικός διάλογος και μια λειτουργούσα βουλή. τίποτα άλλο. Τα εξής τώρα ε, διακυβεύονται στην Αλβανία μια νέα πρόπτικη ε, στη γραμμή των συμπερασμάτων του Συμβουλίου που να βασίζεται στα κριτήρια της Κοπενχάγης, σαφής ταυτοποίηση ε, της νομοδότησης του 2010 ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των 12 προτεραιοτήτων και η ακριβής και αποτελεσματική εφαρμογή από την Αλβανία θα σημάνει έναρξη προταξιακών διαπραγματεύσεων της χώρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι 12 αυτές προτεραιότητες μεταξύ άλλων συμπεριλαμβάνουν και τη βελτίωση ε, των δημοκρατικών θεσμών και του πολιτικού διαλόγου, το κράτος δικαίου και τη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης, την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι 12 αυτές προτεραιότητες είναι τα κριτήρια της Κοπενχάγης δεν είναι απλώς μια άσκηση για τους πολιτικούς. Θα πρέπει να έχουν σαφή ωφέλη, μετρήσιμα για τους πολίτες. Οι Αλβανοί πολιτικοί θα πρέπει επιγόντως ε, να θέσουν στο επίκεντρο ε, του ενδιαφέροντός τους το συμφέρον του αλβανικού λαού. Θα πρέπει να υπάρξει ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για να αντιμετωπίσει τις σημερινές πολιτικές προκλήσεις στην Αλβανία. Για το λόγο αυτό, απίφθηνα επιστολή στον Πρωθυπουργό κύριο Μπερίσα ε, μία εβδομάδα πριν τις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου όπου έθετα ένα χρονοδιάγραμμα, ένα οδικό χάρτη ε, που βασιζόταν σε αυτές τις 12 ακριβώς προτεραιότητες για να βοηθηθεί η Αλβανία να φύγει, να ξεφύγει από το σημερινό διέξοδο. Όλοι θυμόμαστε ε, τις τραγικές εξελίξεις που ακολούθησαν. Δεν είναι πολύ αργά ακόμα. Υπάρχουν σαφή μηνύματα και μία αντιστρεπτά ότι ε, ε, υπάρχει βούληση να ξεπεραστεί το πολιτικό διέξοδο και η πρόσφατη κρίση. Σε τέτοια περίπτωση θα ανταποκριθούμε θετικά. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ε, ζωτικό ρόλο να διαδραματίσει εκεί. Εσείς ως πολιτικοί μπορείτε να στείλετε σαφές μήνυμα σε πολιτικούς. Ένα σαφές ενωμένο μήνυμα από το Κοινοβούλιο και όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση με την προηθυμία μας να βοηθήσουμε να ε, βοηθήσουμε όλους τους Αλβανούς να σκεφτούν ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος δράσης. το με τις ευκαιρίες, κύριε Πρόεδρε και αγαπητοί βουλευτές, για να απευθύνω έκκληση στον Πρωθυπουργό της Αλβανίας, τον κύριο Μπερίσα, να δημιουργήσει ε, πραγματικά ένα πολιτικό περιβάλλον στην Αλβανία που να συμπεριλαμβάνει και όλες τις πολιτικές δυνάμεις και την κοινωνία των πολιτών και τις οργανώσεις και ε, όλοι αυτοί θα ε, επωφεληθούν από την ευρωπαϊκή τους προοπτική. Θέλω να καλέσω και τον ηγέτη του Σοσιαλιστικού Κόμματος, τον κύριο Ράμα, να διαβεβαιώσει ότι το κόμμα του είναι μια επικοδομητική αντιπολίτευση, μια αντιπολίτευση που ε, εποφελείται, αλλά καταλαβαίνει και ποιες είναι οι ευθύνε σε ένα τέτοιο πολιτικό περιβάλλον που να συμπεριλαμβάνει όλες τις πολιτικές δυνάμεις που επιθυμούμε να επικρατήσει στην Αλβανία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Και τώρα θα ακούσουμε τους εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων. Πρώτα, εκ μέρους του Λαϊκού Κόμματος, το λόγο έχει ο Μιχαήλ Γκάλερ. Για δύο λεπτά. Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Επίτροπε, καταρχήν ε, σας ευχαριστούμε πολύ για ε, τα ξεκάθαρα λόγια σας που νομίζω πέτυχαν το στόχο τους. Θεωρώ ότι για να υπάρξει ε, Δρόμο τη Ευρωπαϊκή Ένωση προ την, της Αλβανίας την Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να υπάρχουν δημοκρατικοί θεσμοί. Το Κοινοβούλιο είναι ο χώρο εκείνο όπου πρέπει να λαμβάνει η χώρα η δημοκρατική αντιπαράθεση ε, και γι' αυτό οι πολίτε εκλέγουν τη Βουλή. Ε, το Κοινοβούλιο δεν μπορεί να αντικατασταθεί από τους δρόμου και σίγουρα όχι όπω το προσπάθησε ο κύριο Ράμα στις 21 Ιανουαρίου. Καλό λοιπόν το Σοσιαλιστικό Κόμμα να συνεργαστεί χωρί περιορισμού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εκεί να παρουσιάσει τι πολιτικέ. Σε εναλλακτικές λύσεις. Δεν πρέπει πλέον να αμφισβητείτε το εκλογικό αποτέλεσμα. Η αντιπολίτευση πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της ε, στο Κοινοβούλιο και πρέπει να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία για να συνεργαστεί στην ε, Κοινοβουλευτική Εξεταστική Επιτροπή να καταθέσει προτάσεις για το μέλλον. Υπάρχουν οι προτάσεις του ΟΣΑ για τη βελτίωση των συνθηκών πλαίσιο για τις εκλογές. Εξίσου είναι σημαντικό να συνεργαστούν οι σοσιαλιστές και από ό,τι άκουσα ο κύριος Ράμα εδώ στο Στρασβούργο διαβεβαίωσε ότι θα συμμετάσχει στις, ε, στις δημοτικές εκλογές ε, που θα λάβουν χώρα σύντομα. Ελπίζω λοιπόν ο κύριος Ράμα να ακούσει ε, τις καλές συμβουλές που πήρε εδώ τόσο από τους σοσιαλιστές συντρόφους του αλλά και από εκπροσώπους άλλων πολιτικών ομάδων και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι πολλοί από τη δική μας την πολιτική ομάδα δραστηριοποιούνται για την Αλβανία και ως εκ τούτου αυτή η ε, ευρύτερη προσέγγιση που πρότεινε ο κύριος Επίτροπος που θα συμπεριλαμβάνει όλους ε, στηρίζεται από πολλούς. Με τον τρόπο αυτό θεωρώ ότι όλοι μας ε, συμβάλλουμε έτσι ώστε η Αλβανία να χαράξει ένα αίσιο μέλλον. εκ μέρους των σοσιαλιστών και δημοκρατών το λόγο έχει για δύο λεπτά ο κύριος Ανδριάς Σεβερίν. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε τη σημερινή κατάσταση στην ε, Αλβανία ως αδιέξοδο. Μερικές φορές ε, ήρεμη, μερικές φορές ε, κλιμακούμενη, αλλά δεν έχει τέρμα αυτή η κατάσταση. Είχαμε ψήφισμα το περασμένο χρόνο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο, ζητώντα από όλου του πολιτικού φορεί να διαπραγματευτούν μια πολιτική λύση για να εξέλθουν από την κρίση και να καταλήξουν σε μια ελάχιστη εθνική συνένεση. Δυστυχώ αγνοήθηκε το ψήφισμα αυτό και από τι πολιτικέ δυνάμει, αλλά ιδιαίτερα από την αλβανική κυβέρνηση. Επίσης, οι συστάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και του Συμβουλίου αγνοήθηκαν, έχουν παραγωνιστεί πλήρως από την Αλβανία. Είναι απαράδεκτο η, η άσκηση του δικαιώματος ε, διαμαρτυρίας ε, και έκφραση λόγου μιας χώρας που μαστίζεται από τη διαφθορά να χαρακτηρίζεται ως πραξικοπηματική. Είναι απαράδεκτο τα θεσμικά όργανα της Αλβανίας, ο Πρωθυπουργός ή η, η δικαιοσύνη να υπονομεύονται από δηλώσεις της κυβέρνησης. Είναι απαράδεκτο άνθρωποι που πυροβολούν κατά τον, το αμάχο πληθυσμού και των άοπλων διαδηλωτών να αποκαλούνται εθνικοί ήρωες. Ε, θα γίνουν σύντομα ε, δημοτικές εκλογές στην Αλβανία και θα είναι η λιδία λίθος για όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Ζητώ από τον Επίτροπο Φίλε και τον ε, κ. Βάιτσεκ να κάνουν ό,τι μπορούν για να εξασφαλίσουν διεθνή ενίσχυση αλλά και παρακολούθηση των εκλογών αυτών στην Αλβανία προκειμένου να διεξαχθούν όντω ελεύθερε και δίκαιε εκλογέ και τουλάχιστον να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε κατά πόσο θα είναι τέτοιε. Είμαστε υπέρ τη προσέγγιση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και του Επιτρόπου Φίλε. Υποστηρίζουμε τη δράση του κ. Λάιτσακ και θα πρέπει να παροτρύνουμε όλε τι πολιτικέ δυνάμει Αλβανία να φέρουν σε πέρα σε αυτή την κρίση. Γιατί η εναλλακτική λύση θα είναι η απομόνωση τη Αλβανία. Κάτι τέτοιο θα διακυβεύσει την ενταξιακή της προοπτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστούμε κύριε Σεβερή. Το λόγο τώρα έχει εκ μέρους των φιλελευθέρων και δημοκρατών η κυρία Σάκη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και μέρα σήμερα για την Αλβανία. Μίλησα με εκπροσώπους των δύο βασικών πολιτικών κομμάτων εκεί και του ζήτησα να δώσουν ιδέες και να ανταλλάξουν απόψεις για το πώς θα προχωρήσει η χώρα και πώς θα σπάσει το πολιτικό αδιέξοδο για να αντιμετωπίσουν προβλήματα που αφορούν πολίτε κατά πολέμηση τη διαφθοράς, του οργανωμένου εγκλήματος, δημιουργία απασχόληση και ευκαιριών για τη νέα γενιά. Κανένα από αυτού δεν μου έδωσε απάντηση. Αυτό που τους ενδιέφερε να παίξουν αυτό το παιχνίδι. Ε, το πολιτικό κατεστημένο στην Αλβανία είναι απασχολημένο περισσότερο με τον εαυτό του παρά με το λαό του. Πρόεδρε, δεν χρειάζεται να σας πω πόσο δύσκολο είναι για μας να πείσουμε τους ψηφοφόρους μας να μας ακολουθήσουν όταν ε, ζητούμε διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρά τις αντιστάσεις, η ομάδα μας θέλει τα Δυτικά Βαλκάνια να αποτελέσουν ε, τμήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κοινότητα αξιών η Ευρωπαϊκή Ένωση που άφησε ε, πίσω τις διαιρέσεις του παρελθόντος και επέλεξε ένα μέλλον. Θα πρέπει να καλέσουμε τι αλβανικές αρχές να κάνουν το ίδιο και να μην ασφικτιούν από τις σκιέ του παρελθόντος αλλά να διαβούν προς το φως του μέλλοντος. Είναι δική του ευθύνη πρώτα απ' όλα να φροντίσουν για την εφημερία των πολιτών του για την ευημερία των πολιτών τους και να μην τους ανεθούν το ευρωπαϊκό μέλλον. Γιατί η, πολιτική κρίση δεν βοηθάει την πρόοδο. Νέες εκλογές θα γίνουν το Μάιο, ε, γίνονται οι προετοιμασίες τώρα και θα πρέπει να υποστηριχθούν από όλα τα πολιτικά κόμματα και χαίρομαι για την πρόταση να ε, βοηθήσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση για να γίνουν γνήσιες και ελεύθερες εκλογές, ανώθευτες. Η δημοκρατία όμως είναι μακράς πνοής και δεν είναι απλώς ένας άνθρωπος μια ψήφος. Σημαίνει θεσμούς που να λειτουργούν κράτους δικαίου και σεβασμό για τις μειονότητες. Η δημοκρατία δεν είναι ότι ε, ο νικητής θα παίρνει όλα. Χρειάζεται σκληρή δουλειά και αμοιβαία δέσμευση. Και η μεταρρύθμιση ε, στην Αλβανία θα πρέπει να συνεχιστεί όπως και η δέσμευσή τους προς την ευρωπαϊκή προοπτική. Ευχαριστώ ο Πρόεδρος. Και τώρα το λόγο έχει εξ ονόματος των Πρασίνων και της Ελεύθερης Ευρωπαϊκής Συμμαχίας η κυρία Μαρία Κορνέλισεν για 4,5 λεπτά. Πρόεδρε, η κρίση στην Αλβανία δεν είναι τίποτα καινούριο. Ούτε άρχισε το Γενάρη με τη βία που ξέσπασε κατά των διαδηλωτών. Ούτε το 2009 άρχισε όταν το Σοσιαλιστικό Κόμμα μποϊκόταρε τη Βουλή μετά τις ε, ε, εκλογές. Η κρίση είναι κρίση πολιτικής κουλτούρας, πολιτικού πολιτισμού. Ε, μποϊκοτάζ, απεργία πείνας, διαδηλώσεις είναι συνηθισμένα εργαλεία στην αλβανική πολιτική. Πολιτική διορισμή, διαφθορά και χειραγώγηση του τύπου επίσης. Αυτά απέχουν πάρα πολύ από την πολιτική που εμείς επιθυμούσαμε για μια χώρα που έχει πάρει το δρόμο της ένταξης. Εγώ ε, ε, εύχομαι στους πολίτες της Αλβανίας να έχουν υπεύθυνη κυβέρνηση και υπεύθυνη βουλή με πολιτικούς που βάζουν πάνω από το δικό του συμφέρον και τη δική τους τιμή ε, το συμφέρον του λαού. Θα πρέπει να προχωρήσουν και οι δύο πλευρές, να προσεγγιστούν. Η κυβέρνηση φέρει ιδιαίτερη ευθύνη. Η κυβέρνηση έχει το μονοπόλιο της βίας και η κυβέρνηση έχει ιδιαίτερη ευθύνη να είναι υπερκομματική και να κάνει αυτό που πρέπει για το λαό της. Από την κυβέρνηση αυτή θα πρέπει να περιμένουμε να κάνει ό,τι μπορεί ε, ε, να αποτρέψει φαινόμενα τύπου Ιανουαρίου να επαναληφθούν. Θα πρέπει όλοι να βοηθήσουμε και να πιέσουμε για μια ανεξάρτητη διερεύνηση. Το θέμα της διαφθοράς ε, επίσης πρέπει να αντιμετωπιστεί και να γίνει ευρεία κοινοβουλευτική συζήτηση. Ευθύνη όμως έχει και αντιπολίτευση και η αντιπολίτευση θα πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί για να ε, αποτρέψει η επανάληψη της βίας του Ιανουαρίου ε, για να βοηθήσει να γίνουν σωστές και δίκαιες και γνήσιες εκλογές για να συμμετέχει και στις εκλογές και στην κοινοβουλευτική συζήτηση και επί της ουσίας η ουσία είναι ότι υπάρχει τεράστια ανεργία ας πούμε πώς θα τα κάνουμε τα κόμματα να πάνε αυτή την κατεύθυνση ο Επίτροπος, ο φίλε, τον Νοέμβριο ε, έστειλε τον μπαλάκι στην πλευρά της Αλβανίας και είπε δεν θα υπάρξει επόμενο βήμα πριν ε, κάνετε ε, αυτό που πρέπει. Δυστυχώς αυτό δεν οδήγησε σε αλλαγή. Τώρα ελπίζω με τον κύριο Λάιτσεκ να βοηθήσει να γίνει αυτή η αλλαγή η καμπή και να έρθουν κοντά τα κόμματα. Ελπίδα έχω, αλλά δεν έχω πολύ μεγάλη πίστη ότι θα γίνει αυτό. Μήπως θα πρέπει να σκεφτούμε τίποτα κυρώσεις, να είναι σαφές ότι ε, αν αποτύχουν διαπραγματεύσεις μεταξύ των κομμάτων, αυτό θα έχει και κυρώσεις. Και θα πρέπει να φτάνει και να πλήττει και τους πολιτικούς ηγέτες, όχι το λαό. Άκουσα στους διαδρόμους ότι γίνεται λόγος για κατάργηση θεώρησης διαβατηρίων. Ε, και δεν θα πρέπει τα θέματα ε, αυτά να φύγουν τους πολίτες, επαναλαμβάνω, τους ηγέτες. Κάτι άλλο. Ε, ε, υπάρχουν οι πόροι του πρωταξιακού μέσου ΙΠΑ. Δεν μπορούμε να αφαιρέσουμε την αρμοδιότητα της διαχείρισής του από την Αλβανία και να την έχουμε εμείς. Ως μεσοποίησης. Να είναι υποκειδαιμονία η κυβέρνηση. Ιδού μια κύρωση που δεν πλήττει τους πολίτες αλλά τους πολιτικούς. Θα πρέπει κάπως να οδηγηθούν ε, σε συνεννόηση, σε διάλογο, σε συμβιβασμούς ε, τα κόμματα. Ελπίζω να πετύχει ο κύριος Λάισεκ προς το συμφέρον του αλπαλικού λαού. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα το λόγο έχει εξ ονόματος ε, της ομάδας των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών ο κύριος Τσάλτς Τάνοκ. Για δύο μισή λεπτά, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, εάν η Αλβανία επιθυμεί να σημειώσει πρόοδο προ τον στόχο που είναι η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι πολιτικοί, της πολιτική ηγέτε πρέπει να συμμετάσχουν πολύ πιο όρημα και επικοδομητικά. Η βία του περασμένου μήνα ε, υπενθύμησε το κληροδότημα τη Αλβανία στην πολιτική. Το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει ίσω να αναθεωρήσουν την απόφασή του που έλαβαν πέρυσι να ε, δώσουν την δυνατότητα να ταξιδεύουν οι πολιτέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρί ε, ε, Βεβαίω, ε, ε, αν δεν υπάρξουν επενδύσεις στη χώρα θα υπάρξει μεγαλύτερη μετανάστευση και αυτό υπογραμμίζει το γεγονό ότι η Αλβανία εξακολουθεί να μην ανταποκρίνεται στις προσδοκίες Ευρωπαϊκή Ένωση. Το οργανωμένο έγκλημα και η διαφθορά εξακολουθούν να διαδίδονται, ε, υπάρχουν όλοι χειρισμοί. Ο Πρωθυπουργό κ. Μπερίσα μάλιστα ε, παρενέβη στην, στον Γενικό Εισαγγελέα όταν συνελήφθησαν οι αστυνομικοί και πολλοί έλεγαν ότι θα υπάρξει πραξικό δεν υπάρχουν ελευθερίε, πολύ λίγε είναι αυτέ, ε, αλλά και το Σοσιαλιστικό Κόμμα του κ. Ράμα να μποϊκοτάρει το Κοινοβούλιο, ε, διότι υποτίθεται ότι υπάρχουν, ε, υπήρξε εκλογική νοθεία. Αυτό αποδυναμώνει περαιτέρω την Αλβανία. Η Αλβανία δεν μπορεί να εφαρμόζει τι μεταρρυθμίσει για να αποκτήσει ξανά την εμπιστοσύνη τη Ευρωπαϊκή Ένωση με τα γεγονότα που υπάρχουν. Αυτή λοιπόν η αστάθεια καλεί και το ΝΑΤΟ να αναθεωρήσει και αυτό την πολιτική του τη διεύρυνση. Η Αλβανία μπήκε στο ΝΑΤΟ πριν από δύο περίπου χρόνια χρόνια και τώρα οι ηγέτε του ΝΑΤΟ θα πρέπει να ερωτηθούν ε, τα πόσα μήπω τι έδωσαν πολύ εύκολα και γρήγορα αυτή την ένταξη. Με απασχολεί η αστάθεια τη Αλβανία. και επίση ε, είμαι και πολύ σκεπτικό όσον αφορά τι στρατηγικέ προτεραιότητε τη Αλβανία. Η Αλβανία είναι πλήρε τη τη οργάνωση ε, Συνοργάνωση ε, και Συνδιάσκεψη και έτσι προάγει τα συμφέροντα των μελών. Όλοι ψηφίζουν ενσώματοι για τα ανθρώπινα δικαιώματα και θέματα πολιτική. Η Αλβανία και η Τουρκία έχουν υπογράψει το χάρτη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, στις ε, μουσουλμανικές χώρες. Η Αλβανία όπως και η Τουρκία θα πρέπει να αποφασίσουν αν θέλουν να προσχωρήσουν στις δυτικές αξίες ή στη Σαρία ε, που το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εδώ στο Στρασβούργο έχει κρίνει ότι είναι ασυμβίβαστο με τις ευρωπαϊκές αξίες. Κατά την άποψή μου λοιπόν η Αλβανία επειδή είναι μέλος του ΟΣΑ μόνο κατόνομα η Αλβανία Αλβανία ε, στην πρακτική βέβαια είναι μια λαϊκή χώρα και οι Αλβανοί, οι ηγέτες ε, της Αλβανίας από ό,τι φαίνεται μπήκαν στον ΟΣΑ για να προσελκύσουν τα χρήματα της Μέσης Ανατολής και όχι για θρησκευτικούς λόγους. Ελπίζω λοιπόν όλα αυτά να αλλάξουν στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο τώρα έχει ο κύριος Χουντής παρακαλώ για τρία λεπτά. Εξ ονόματος της ομάδας του. Παρακαλώ κύριε πρόεδρε αγαπητοί συνάδελφοι κύριε επίτροπε είχα την ελπίδα ότι ενάμιση χρόνο μετά τις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές στην αλβανία θα είχε τελειώσει θα είχε λυθεί το πολιτικό αδιέξοδο. είχα την ελπίδα ότι μετά τις συστάσεις με το ψήφισμα του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου θα λαμβάνονταν υπόψη αυτά που λέγαμε. είχα την πεποίθηση ότι η προσδοκία για ευρωπαϊκή ένταξη της αλβανίας θα αποτελούσε ισχυρό κίνητρο εφόσον το επιθυμούν οι αλβανοί πολίτε, για τη λύση όχι μόνο του πολιτικού προβλήματο, αλλά και των οικονομικών κοινωνικών και δημοκρατικών ε, προβλημάτων. Δυστυχώ, το αδιέξοδο συνεχίζεται. το ποιο έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη πιστεύω αγαπητοί συνάδελφοι δεν είναι δικό μα έργο θα το κρίνει ο Αλβανικό λαό. Δυστυχώ όμω τα πράγματα έχουν γίνει χειρότερα. εκφράζω για άλλη μια φορά τη θλίψη μου για τα θύματα τη διαδήλωση τη 21 η του Ιανουαρίου. Είμαστε αντίθετοι στην κλιμάκωση τη βία, ζητούμε να σταματήσει η καταστολή, να γίνεται σεβασμό των ανθρωπίνων και των δημοκρατικών δικαιωμάτων και να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι. Όμω δεν σα κρύβω ότι είμαι ανήσυχο εν ώψη των επικείμενων δημοτικών ε, εκλογών, τοπικών εκλογών πρέπει, του Μαΐου. Πρέπει οπωσδήποτε, εδώ πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, να γίνουν ε, και να διασφαλιστούν όλες οι αναγκαίες εγγυήσει ούτω ώστε να γίνουν ομαλά. είναι θετικό και πρέπει να πιέσουμε να μετέχουν όλε οι πολιτικέ δυνάμει σε αυτή την εκλογική διαδικασία να διεξαχθούν αυτέ οι εκλογέ είναι πάρα πολύ κρίσιμο με του διεθνού κανόνε των αδιάβλητων και δημοκρατικών εκλογών. αγαπητοί συνάδελφοι πιστεύω πω η βοήθεια η δική μα η βοήθεια του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και τη ευρωπαϊκή ένωση γενικά και συμφωνώ με την τοποθέτηση του κ. φούλε πρέπει να είναι επικουρική πρέπει να είναι βοηθητική και προφανώς δεν πρέπει να χαρακτηρίζεται από κομματική συγγένεια και από πολιτικές φιλίες επιτρέψτε μου την έκφραση. δεν θα δώσουμε εμείς τη λύση αγαπητοί συνάδελφοι στην αλβανική κοινωνία και στο αλβανικό πρόβλημα. αυτό πρέπει να είναι υπόθεση του αλβανικού λαού των αλβανικών πολιτικών δυνάμεων. δεν συμφωνώ με σκέψεις που ακούγονται για απειλές λήψης μέτρων όταν τα περισσότερα από αυτά ε, που ακούγονται είναι μέτρα που θα είναι σε βάρο των αλβανών πολιτών και δεν νομίζω ότι θα έχουμε κανένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. πιστεύω ότι μέσα από τα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα στο πλαίσιο των σχέσεων μια χώρα που είναι στον προθάλαμο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, εκεί μπορούμε να ασκήσουμε τη μεγαλύτερη επιρροή λέγοντα ότι όλε αυτέ οι διαδικασίε δυστυχώ καθυστερούν αυτή την ενταξιακή προοπτική και πρέπει να επισημάνουμε ότι το αδιέξοδο θα έρθει αγαπητοί συνάδελφοι μόνο με υπεύθυνη πολιτική στάση των πολιτικών ηγετών με τη λογική του διαλόγου του διαλόγου του πολιτικού διαλόγου και της ε, λογικής και όχι με πρακτικές και συμπεριφορές που όπως υπόθηκε ο νικητής τα παίρνει όλα. πιστεύω ότι αν επιμείνουν οι πολιτικοί ηγέτες της αλβανίας σε αυτή την πρακτική και σε αυτή τη λογική το αδιέξοδο θα ενταθεί και η κρίση θα βαθύνει και έτσι δεν θα μπορέσει να αντιμετωπίσει η χώρα αυτή σοβαρά προβλήματα εκτός από το πολιτικό πρόβλημα προβλήματα που θα προκύψουν και προκύπτουν από την οικονομική κρίση η οποία πλήττει τις γειτονικές χώρες την ιταλία και την ελλάδα όπου τα εμβάσματα από αυτές τις χώρες βοηθούσαν ως ένα βαθμό την οικονομική κατάσταση της αλβανίας. επομένως η άρση του πολιτικού αδιεξόδου η πολιτική υπευθυνότητα ο πολιτικός διάλογος είναι αυτό που πρέπει να οδηγήσει τους πολιτικές ηγέτες να δώσουν γρήγορα λύση στο πρόβλημα που έχει η αλβανία. ευχαριστώ πολύ. Thank Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ. Και τώρα το λόγο έχει ο κύριος Μπέλτερ. Δυόμιση λεπτά εξ ονόματος της ομάδας της Ευρώπης Ελευθερίας και Δημοκρατίας. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ως δημοσιογράφος στη δεκαετία του 90 επισκέφθηκα πολλές φορές στην Αλβανία και ε, συνέχεια με εντυπωσίασαν οι νέοι, τα λαντούχοι νέοι. Μια χώρα με τέτοια νεολαία θα έπρεπε να έχει μέλλον. Πέρσι το καλοκαίρι και πάλι ενθαρρύνθηκα ε, ε, όταν πήγα στον Αυλώνα και ενημερώθηκα για την ευρωπαϊκή προοπτική. Και μάλιστα εντυπωσιάστηκα από δύο νέους 30 ετών ε, που ε, εργάζονται στη χώρα που δεν έφυγαν θα μπορούσαν να είχαν φύγει. Και ήταν και ένας εκπρόσωπος του κλήρου και ένας εκπρόσωπος του λαού ε, και μας είπαν ότι η Ευρώπη δεν θα πρέπει να αφήσει τους πολιτικούς μας ηγέτες στη μοίρα τους. Η Ευρώπη θα πρέπει να βοηθήσει να φέρουν τα δύο κόμματα σε διαπραγματεύσεις, το δεξιό κόμμα και το σοσιαλιστικό. Κύριε Επίτροπε, ε, ε, ομολογώ ότι αυτό είναι πιο εύκολο να το λες παρά να το κάνεις. Δεν θα πρέπει όμως να χάσουμε την ελπίδα μας και γιατί έχουν αναποθέσει στα δικά μας χέρια την ελπίδα τους πολλοί Αλβανοί νέοι. Πραγματικά ε, θέλω να σας βοηθήσω αυτή την προσπάθεια, σας με κάθε επιτυχία και κάτι άλλο που δεν είναι ίσονο σημασία για την Αλβανία. Στα Τύρανα μου επέσαν την προσοχή ε, στο εξή γεγονός. Πέρυσι Πολλές Αλβανές γυναίκες και κορίτσια διακινήθηκαν στην Ευρώπη παράνομα για να καταλήξουν στην πορνεία. Πώς θα το σταματήσετε αυτό, τι μέσα έχουμε στη διάθεσή μας. Γιατί ανθεί αυτό το εμπόριο στην Αλβανία. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τέλος ε, για τους ανεξάρτητους ο κύριος Μπιλοκόβατς για ένα λεπτό. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Από τις εκλογές του 2009 η πολιτική ζωή στην Αλβανία έχει περιέλθει σε αδιέξοδο. Το Κοινοβούλιο και τα θεσμικά όργανα δεν φαίνεται να λειτουργούν. Το γεγονός ότι οι σοσιαλιστές κατηγορούν την κυβέρνηση για ανοθεία και δεδομένου του ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήθελε να γίνουν πρόορες εκλογές και το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός ο κύριος Μπερίσα δεν θέλει να απομακρυνθεί από τη θέση του ε, και κατηγορεί την αντιπολίτευση για βία όλα αυτά μου δίνουν την εντύπωση πως οι διαπραγματεύσεις θα αποτύχουν. χώρες ε, που θέλουν να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αντιμετωπίσουν το οργανωμένο έγκλημα. Αυτό δεν είναι σημαντικό μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και για τις ίδιες χώρες. Βοηθούν και την, βοηθά και την εικόνα της χώρας ε, κάτι τέτοιο. Οπότε για να βελτιωθεί η κατάσταση στις χώρες αυτές είναι σημαντικό να αποκατασταθούν οι δημοκρατικοί θεσμοί σε αυτές τις ε, χώρες. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τώρα το λόγο έχει ο κύριος Εντουαρντ Κούκαν για δύο λεπτά για το ΕΛΚ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, συνάδελφοι. Η πολιτική κρίση στην Αλβανία έχει κρατήσει πάρα πολύ. Ναι, δεν είναι αδιέξοδο. Είναι μια παρατεταμένη πολιτική κρίση. Βλάπτει την εικόνα της χώρας, τους πολίτες τους και τις φιλοδοξίες τους για το ευρωπαϊκό τους μέλλον. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε σε αυτή την πολιτική κρίση και τις εντάσεις να συνεχιστούν. Αυτό το οποίο χρειαζόμαστε τώρα είναι να στείλουμε ένα κοινό μήνυμα πώς θέλουμε η Αλβανία να είναι υποψήφια χώρα. Αλλά οι πολιτικοί ηγέτες και από τις δύο πλευρές πρέπει να επιδείξουν την ε, βούληση να λύνουν τα πολιτικά προβλήματα σεβόμενοι το κράτος δικαίου, το Σύνταγμα και επί τη βάση δημοκρατικών θεσμών. Προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε εδώ και καιρό να βρεθεί μια λύση στο πρόγραμμα χωρίς από το αποτέλεσμα. Καταδικάζουμε την βία στους δρόμους των τυράννων ε, στις ε, διαδηλώσεις της 21ης Ιανουαρίου. Γεγονότα που κόστησαν τη ζωή τεσσάρων ανθρώπων, τα οποία πρέπει να ερευνηθούν. Η Αλβανία αναμένει τις ε, τοπικές εκλογές του Μαΐου, οπότε θα έχουμε άλλον έναν έλεγχο για δημοκρατία στη χώρα. Και πάλι λοιπόν θα πρέπει να δώσουν εγγυήσει οι πολιτικές δυνάμεις για το ότι οι εκλογές δεν θα σημάνουν περαιτέρω ετάσεις και παράταση της κρίσης. Συμπερασματικά, κύριε Πρόεδρε, θέλω να τονίσω τη σημασία των πολιτικών μηνυμάτων και προτάσεων που περιέχονται στον λόγο του Επιτρόπου Φίλε στην αρχή αυτής της συζήτησης. Η καλύτερη θετική συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπ' αυτές τις συνθήκες είναι να ρίξει όλο του το βάρος πίσω από αυτές τις προτάσεις και να στείλει ένα σαφές κοινό μήνυμα στα αλβανικά κόμματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος ε, Χάνες Φόμποντα έχει τον λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο, τον κύριο Φιούλε για αυτά τα οποία είπε, σαφώς. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Λάιτσεκ για την δική του εμπλοκή που τους τελευταίους μήνες. Είναι συνηθισμένος να αντιμετωπίζει και να λύνει αγκαθόδη προβλήματα και νομίζω πως ε, υπάρχει μια κοινή διάθεση εδώ πέρα που προέκυψε από αυτή τη συζήτηση και βλέπω πως ε, και οι δυο σας ε, είστε κάπως συγκρατημένοι. Κοιτάξτε, εγώ ομολογώ πως είμαι κάπως επιφυλακτικός για την ε, συζήτηση, γιατί το χειρότερο είναι να ανταλλάσσουμε εμείς εδώ πέρα κατηγορίες, όπως ακριβώς κάνει στην Αλβανία η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση. Θα πρέπει λοιπόν και οι δύο πλευρές, και η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση, να τηρήσουν αυτό το που έχουν πει για να βρεθεί μια διέξοδος από την λύση. Γιατί, όπως είπε και ο κύριος ε, Μπέλτερ, και εγώ είχα πάει όταν έπισε το καθεστώς Χότζα στην Αλβανία και είχα συγκινηθεί από το, την ατμόσφαιρα που επικρατούσε, από το πόσο ικανοποιημένοι ήταν οι νέοι, από το τι περίμεναν και όταν βλέπουμε το τι δεν έγινε τελικά, η απογοήτευση είναι μεγάλη. Και η πολιτική τάξη στην Αλβανία δεν είναι ικανή να ικανοποιήσει τις επιθυμίες του λαού. Βεβαίω υπάρχουν οι πολιτικές συγγένειές μας, οι προσωπικές φιλίες, αλλά το αποφασιστικό είναι να πούμε και στις δύο πλευρές καθίστε μαζί να τα βρείτε και προσπαθήστε τουλάχιστον οι δημοτικές εκλογές να είναι διαφανείς. Και πρέπει να απευθύνουμε πρόκληση και οι δύο να είναι έτοιμοι. Αυτό το οποίο διαπίστωσε ο κύριος Σοντή, να γίνουν τα απαραίτητα για αυτέ τι εκλογέ, είτε μέσω νομοθεσία, είτε μέσω εφαρμογή νομοθεσία για να είναι σωστέ αυτές οι εκλογέ. και θα πρέπει να στείλουμε όσο δυνατόν περισσότερου ε, εκλογικούς, παρατηρητέ, παρατηρητές παρά το ότι είναι δημοτικές εκλογές γιατί μπορούν να αποτελέσουν την αφετηρία ενός νέου κλίματος στην Αλβανία. Η Αλβανία σε αυτό συμφωνούν όλοι, εάν δεν αλλάξει τίποτα θα απομονωθεί. Δεν θέλουμε να απομονωθεί η Αλβανία, θέλουμε να μπει σε έναν δρόμο προς την Ευρώπη. Ευχαριστώ. Και τώρα ο κύριο Στάνιμιρ Ιλτσεφ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Να ξεκινήσω δηλώνοντας πως η αλβανική κοινωνία, ο αλβανικός λαός είναι ιδιόμορφοι και σας παρακαλώ πολύ μην με παρεξηγήσετε, αλλά έχουν μια πολύ συγκεκριμένη πολιτική κληρονομιά, παραδόσεις, πολιτισμό και μέχρι σήμερα έχουν διατηρήσει αυτές τις ιδιομορφίες. Ο, εθνικός τους χαρακτή, ο χαρακτήρας τους εθνικά είναι ιδιόμορφος και ο τρόπος που αντιμετωπίζουν τις πολιτικές διαδικασίες είναι επίσης ιδιόμορφος. Πρέπει να είμαστε λοιπόν εμείς ευέλικτοι και δημιουργικοί, εφευρετικοί θα ήθελα να πω, στην αντιμετώπιση τους και να μην παραμείνουμε μόνο σε επαφή με τις δύο αντιμαχόμενες πολιτικές πλευρές αλλά και με τους άτυπους ηγέτες της αλβανικής κοινωνίας. Πολλά, πολλά θετικά σχόλια ακούστηκαν εδώ ε, και για την ε, Σαριά και για τις άλλες δημορφίες αλλά εκεί έχουμε τρεις ε, θρησκείες την Ορθοδοξία, ε, τον Καθολικισμό και το Ισλάμ έχουμε εκεί λοιπόν τους θρησκευτικού ηγέτες έχουμε τους ηγέτες της νεολαίας παρακαλώ μην τους αφήσουμε στην άκρη Ευχαριστώ πολύ και θα δώσω το λόγο τώρα στην κυρία Λούνα Τσέκα Έχετε τρία λεπτά Ευχαριστώ Κύριε Πρόεδρε, κύριε Φίλε, κυρίες και κύριοι, και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τους κυρίους ε, Φίλε και Λάιτσα για αυτά τα κάνουν και προσπαθούν να κάνουν για να βρεθεί μια διέξοδος και για τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ξεκινήσει μια διαδικασία στήριξης της Αλβανίας. Θεωρώ πως ε, η σημερινή συζήτηση δεν πρέπει να γίνει καυγά των πολιτικών οικογενειών που συγκρούονται και εντός της Αλβανίας θα ήταν θλιβερό αυτό για το κοινοβούλιο μας και ελπίζω να μην είναι έτσι τα πράγματα. Η θεσμική κρίση της ε, Αλβανίας είναι μια κρίση πολιτικής ε, κουλτούρας. Ε, μιλάμε για λεκτική βία που μεταφράζεται μετά σε βία στους δρόμους όπου πεθαίνουν άνθρωποι. Πρέπει να ερευνηθεί αυτό το περιστατικό και το ποιος θέλει. Αλλά η στάση αυτή της λεκτικής βίας που οδηγεί σε πραγματική βία είναι πραγματικά κάτι το οποίο μπορεί να θέσει εν κινδύνο την ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας. Και όπως είπε ο κύριος Φιούλε, θα πρέπει πραγματικά οι αντιμαχόμενοι στην Αλβανία να αντιληφθούν πως ε, πρέπει να δράσουν προς το συμφέρον του αλβανικού λαού. Και εδώ πέρα αυτό σημαίνει δρόμος προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, μία λύση για την πολιτική κρίση, να καθίσουν σε ένα τραπέζι και να σταματήσουν να κατηγορούν ο ένας τον άλλον και όλο ο άλλος φταίει και να μην ε, βλέπουν πώς μπορούν και οι ίδιοι να συνεισφέρουν κάτι για να αλλάξει η κατάσταση. Αυτό χρειάζεται για Ε, να δούμε τι θα γίνει. Και βέβαια το ποιο ξεκίνησε και το ποιο θέλει δεν είναι πράγματα που γίνονται σε ένα ευρωπαϊκό κράτος. Ο δε κύριος ε, Λάμερ μας ανακοίνωσε πως ε, πράγματι θέλουν και τα δύο κόμματα να λάβουν μέρος στις τοπικές εκλογές. Αυτό είναι κάτι το θετικό και ελπίζω πράγματι να γίνει αποδεκτό και το αποτέλεσμα. Η απελευθέρωση της ε, βίζας ε, και αυτή ε, έτυχε πάρα πολύ μεγάλη υποστήριξη από το Κοινοβούλιο και ελπίζω κύριε Επίτροπε η Κομισιόν να μην σκέφτεται να άρει ξανά την απαλλαγή βίζας των Αλβανών πολιτών ως κύρωση κατά των δύο κομμάτων. Το άλλο ερώτημα είναι ποιες δυνατότητες υπάρχουν εάν δεν συμφωνήσουν οι δύο για να ασκηθεί η πίεση. Μία δυνατότητα, όπως υπόθηκε ήδη, είναι στο πλαίσιο του Ταμείου της Ευρωπαϊκής Εταιρικής Σχέσης να κάνει η Κομισιόν την διαχείριση ή να παγώσει το Ταμείο αυτό, αλλά βεβαίως τότε μόνο ο λαός θα υποφέρει. Οπότε τι προτείνετε για την περίπτωση που δεν θα βρεθεί λύση, κάτι το οποίο δεν ελπίζω. Και τέλος, η έκθεση Μάρτη στο Συμβούλιο της Ευρώπης ε, μίλησε για εμπόριο οργάνων με τη στήριξη για των αλβανικών μυστικών υπηρεσιών. Πώς βλέπετε την ε, διάθεση συνεργασίας ε, της αλβανικής δικαιοσύνης και μυστικών υπηρεσιών εδώ πέρα. Ευχαριστώ. Κύριος Γιάροσλαβ Πάσκα. Για ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Από το 2009 επικρατούει ε, πολιτική ένταση στην Αλβανία λόγω των ε, αποτελεσμάτων των εκλογών οι οποίες θεωρήθηκαν νοθευμένες ε, σοσιαλιστές υπό τον Έντι Ράμα κατηγορούν τον Σαλιμπερίσα για νοθεία αλλά και για το ότι είναι υπεύθυνος για την διαφθορά και την επιδείνωση της κατάστασης ε, στην οποία ζει ο λαός. Οι διαμαρτυρίες της 20 Ιανουαρίου ε, έγιναν με τη συμμετοχή 20.000 ατόμων που ζήτησαν ε, την παρέτηση του Πρωθυπουργού. Επενέβη η αστυνομία με κανόνια νερού, δακρυγόνα και το αποτέλεσμα ήταν τέσσερις νεκροί και πάνω από 150 η δε κτηνοδία της ε, αστυνομίας, της αστυνομικής παρέμβασης είναι πρωτόγνωρη. Σε δημοκρατικές χώρες ε, οι εκλογές ε, κρίνουν το αποτέλεσμα εάν έχει ξεχάσει ο Σαλή Μπερίσα τις ε, βασικές ε, δημοκρατικές αρχές τότε δεν έχει πλέον καμία δουλειά στο αξίωμα το οποίο κατέχει. Εμείς ε, δεν θεωρούμε πως πρέπει να έχουμε δικτατορίσκους στην Ευρώπη που δεν είναι ικανοί να παραδώσουν την εξουσία. Γι' αυτό και θα πρέπει να υποστηρίξουμε τη δημοκρατία στην Αλβανία. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν περιορισμοί χρονικοί. Δεν θα ήθελα να καθυστερήσουμε παραπάνω από όσο έχει προβλεφθεί. Ούτε μου αρέσει να σας διακόπτω όσο έχετε το λόγο, αλλά σας παρακαλώ πολύ να σέβεστε. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Λάιτσεκ, αυτό το οποίο συζητάμε σήμερα δεν ξεκίνησε στις 21 Ιανουαρίου. Γι' αυτό πρέπει να ρωτήσουμε και σας ερωτώ γιατί η Κομισιόν και λοιποί διεθνείς οργανισμοί δεν έζησαν τη φωτιά όταν ξεκίνησε. Δηλαδή στα μέσα του 2009. Οι εκλογές του 2009 ήταν οι καλύτερες μέχρι τώρα και βασίστηκαν σε έναν εκλογικό νόμο το οποίο ακούσατε, ακούσατε, ψηφίστηκε από κοινού από σοσιαλιστές και δημοκράτες. Κάτι το καινούριο στην Αλβανία τότε όλοι οι σοσιαλιστές εκπρόσωποι, οι ΟΝΤΙΡ, εμείς οι ίδιοι είπαμε πως ήταν σωστές οι εκλογές. Και η κυβέρνηση που ακολούθησε ήταν κάτι το καινούριο. Συνεργάστηκαν δύο αντίπαλες ε, δυνάμεις. Το Δημοκρατικό Κόμμα και το μικρότερο Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα. Κάθισαν αυτοί οι δύο εχθροί μαζί για να προχωρήσει η Αλβανία προς τα εμπρός. Είναι στο ΝΑΤΟ, απαλλάχθηκε από τη Βίζα, ακόμα δεν είναι υποψήφια χώρα, αλλά μόλις σχηματίστηκε η κυβέρνηση αποφάσισε η αντιπολίτευση πως δεν ήταν καλές ε, και σωστές οι εκλογές και ζήτησε να ανοίξουν οι κάλπε. κάλπες. Ποιο το κάνει, ποια κυβέρνηση το κάνει αυτό, ούτε στη δική μα ούτε στη δική σα χώρα. Δηλαδή υπάρχει συνταγματικό δικαστήριο και ε, επιτροπή διεξαγωγή εκλογών ή δεν υπάρχει και ξεκίνησαν μετά απεργίε πίνε, αρνήθηκε να συνεργαστεί στο κοινοβούλιο, στην ομοθεσία. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Φταίει κάποιο συγκεκριμένα και πρέπει να το πούμε. Δεν μπορεί να εξισώνουμε συνέχεια του ανθρώπου. Πρέπει να πούμε πού είναι οι δυσκολίε. Αυτό το οποίο αναφέρθηκε ήταν να ανοίξουν οι κάλπες. Δεν γίνεται αυτό γιατί δεν το επιτρέπει το Σύνταγμα. Οπότε τι διαπραγματευόμαστε αν δεν επιτρέπεται. Και μετά είχαμε την κλιμάκωση, είχαμε τέσσερις νεκρούς και καλό είναι το οποίο προσπαθήσατε σήμερα να κάνετε έναν οδικό χάρτη, τέλος πάντων υπερβάλλω λίγο. Και κύριε Λάιτσα και εσείς κύριε Φίλε θα πρέπει να βοηθήσετε τους ανθρώπους αυτής της χώρας για να έχουν ένα καλύτερο μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα το λόγο έχει ο κύριος Βίκτορ Μποστινάρου για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, καλωσορίζω τη δήλωσή σας και θα ήθελα να υπογραμμίσω και την συμβολή του κυρίου Λάτζακ στην προσπάθεια εξέβρεσης λύσεων για να υπερπηδηθεί η δραματική αυτή κατάσταση. Υπάρχουν Διαδηλώσει στην Τινησία και την Αίγυπτο, όπου ο λαός ξεσηκώνεται κατά των δικτατόρων που τελικά αναγκάστηκαν να φύγουν από τις χώρες τους, χωρίς όμως να υπάρξει βία και εκτελέσεις όπως συνέβη στο Τύρανο, όπως είδαμε από τα ΜΜΕ. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό Σαλή Μπερίσα, όπου ε, οι διαμαρτυρόμενοι δεν ήταν παρά υποκινούμενοι από την αντιπολίτευση προσπαθώντας να επιφέρουν ένα πραξικόπημα, ο επικεφαλής ε, των ε, υπηρεσίας ασφάλειας και ο επικεφαλής αστυνομία που όλοι είχαν οριστεί υπό τον Σαλή Μπερίσα, πείτε μου, τι είναι, είναι σοσιαλιστές ή κάτι δεν πάει καλά με τον κύριο Μπερίσα. Θα ήθελα και να αναφέρω κάποιες φράσεις ε, από τον ε, Υφυπουργό Εξωτερικών τον ΗΠΑ, ο οποίος δημοσίως ε, απέριψε το ότι αυτό που συνέβη στις 24 Φεβρουαρίου ήταν πραξικόπημα. Θα πρέπει πραγματικά να είμαστε αποσιωμένοι εδώ και όπως είναι κατηγορηματική η ΙΠΑ και τον ΝΑΤΑ στην προσπάθεια ε, αποστολής βοήθειας στην Αλβανία προκειμένου να επιτευχθεί κάποια λύση κατόπιν διαπραγματεύσεων. Κάνω έκκληση όμως και σε όλους τους συναδέλφους που δίνουν υποστήριξη ανεφόρων στον κύριο Μπερίσα να πάψουν να έχουν αυτή την μονομερή προσέγγιση. Είναι σημαντικό να ασκηθεί πίεση και στις δύο πλευρές και να αναγκάσουμε θέλετε και τις δύο πλευρές να βρουν μια λύση. Μέχρι στιγμής Μόνο η μία πλευρά έχει δείξει κάποια σχετική προθυμία να εφαρμόσει το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τις 12 προτάσεις που αναφέρατε προηγουμένως κύριε Επίτροπε. Ζητώ τώρα από την Επιτροπή να δείξει σταθερότητα και ε, στεναρότητα στην υποστήριξη του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των 12 όρων που αναφέρεται προηγουμένως, λαμβάνοντας υπόψη ότι χωρίς πλήρη συμφωνία και των δύο πλευρών, δηλαδή η, η διαδικασία ευρωπαϊκής ε, ένταξης της Αλβανίας Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να παγώσει όλος καιρό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ και τώρα σε ζητώ, επαναλαμβάνω, ζητώ από όλους να τηρείτε το χρόνο σας, λέει ο Πρόεδρος. Ο κύριος ε, Αντώνιο Κανκιάν για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Σημερίζομαι πλήρως την, τον χάρτη τον οποίο ε, υποβάλλατε και υποδείξατε στην Αλβανία απόψε. Είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι πρόκειται για μια χώρα που έχει ευρωπαϊκή προοπτική. Ω εκ τούτου πρέπει να είναι υποψήφια προς ένταξη. Η, τα θλιβερά γεγονότα της 21ης Ιανουαρίου μας γύρισαν και τα χρόνια πίσω. Είδαμε τις ίδιες σειρές ε, βίας και διαδηλώσεων που, είδαμε που βλέπαμε στη δεκαετία του 90. Πραγματικά ανησυχώ λοιπόν για σχέση με τις πρόσφατες εξελίξεις και τις επιπτώσεις του στο μέλλον της χώρας. Και ο ίδιος μαζί με άλλους συναδέλφους μπόρεσα να θέσω τον τύπο των ήλων τις διάφορες δύσκολες συνθήκες που βιώνει αυτή η χώρα στις τελευταίες επίσκεψή μου του Νοεμβρίου του 2010 ως μέλος της Επιτροπής Νοτιοανατολικής Ευρώπης Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πριν ε, στις 3 και 4 ε, Μαΐου άλλη αποστολή που είχαμε κάνει. Καταφέραμε να κλείσουμε με ένα τελικό ψήφισμα συνεργασία, ε, συμφωνίας. Είναι πιθανόν, αν θέλετε, να μην βρισκόμαστε να μην έχουμε πλήρως ε, επίλυσει διάφορα πραγματικά προβλήματα που είναι η ανεργία, ο πραγματικός δηλαδή κοινωνικός καρκίνος και πέρα από τις άλλες πολιτικές αλχημίες είναι ακριβώς να ξεβρεθεί η συγκεκριμένη ευθύνη η οποία υπάρχει, ποιοι είναι οι υπόλογοι. Είναι απαραίτητο να εγγυηθούμε με κάθε τρόπο να προσπαθήσουμε να υπάρχει μια σύγκληση τουλάχιστον πάνω στο βασικό δίκαιο. Τόσο η πλειοψηφία όσο και η μειοψηφία να συμφωνήσουν από αυτό ώστε οι επόμενες εκλογές να υπάρξει όσο το δυνατόν επικράτηση διαφάνειας και δημοκρατίας. Έχουμε την ευκαιρία σήμερα εν ώψη του ε, 8 Μαΐου που θα συμμετάσχουμε ε, ως παρατηρητές στις δημοτικές εκλογές για το Δήμο των Τυράννων θα είμαστε σε θέση να μετρήσουμε την πραγματική πολιτική δημοκρατία, την πολιτική κατάσταση. Δεν θα πρέπει να κουραζόμαστε πέρα από την πρόοδο που έχει σημειωθεί στις χώρες τελευταία χρόνια, δεν θα πρέπει να κουράζεται η Ευρώπη να συνεχίζει το διάλογο και να συνεργάζεται. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εργασία που θα κάνετε κύριε Επίτροπε, γιατί η παρουσία μας εκεί είναι εξαιρετικά σημαντική. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η κυρία Κοπά, για 1,5 λεπτό. Με ανησυχία παρακολουθούμε τα γεγονότα που διαδραματίζονται στην Αλβανία. Οι δραματικές εξελίξεις στη διαδήλωση που πραγματοποιήθηκε ενάντια στη διαφθορά, με θύματα μετά από συγκρούσεις με δυνάμεις ασφάλειας, πρέπει να καταδικαστούν ρητά. Η συνεχιζόμενη πολιτική κρίση εγκυμονεί πολύ σοβαρούς κινδύνους για τη σταθερότητα στη χώρα όλοι έχουν μερίδιο ευθυνών όμως η εκλεγμένη κυβέρνηση οφείλει να λάβει το μήνυμα που στέλνει ο λαός ότι η χώρα χρειάζεται χρηστή διακυβέρνηση. η δημιουργία κράτους δικαίου με πάταξη της διαφθοράς έπρεπε να είναι στις προτεραιότητες της αλβανικής κυβέρνησης. ο λαός έχει δικαίωμα να διαδηλώνει μέσα στο πλαίσιο της νομιμότητας όταν θεωρεί ότι οι πράξεις της κυβέρνησης στρέφονται σε βάρος του η ευρωπαϊκή ένωση πρέπει να συμβάλλει με κάθε τρόπο ώστε να επικρατήσει ψυχραιμία και σύνεση. στη διαδικασία αυτή όλοι πρέπει να είμαστε παρόντες. καλώ του συναδέλφου του λαϊκού κόμματος να μην παραβλέπουν τις βαρύτατες ευθύνες της κυβέρνησης και να κατηγορούν αποκλειστικά και μόνο την αντιπολίτευση για την πολιτική κρίση. στην παρούσα φάση είναι θεωρώ απαραίτητο να ξαναρχίσει ο πολιτικός διάλογος και να βρεθεί μια λύση μέσα από τι διαδικασίες που ορίζει το σύνταγμα και οι νόμοι. ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τελευταίος αγορητής ο κύριος Μπουσοτήλ, δύο λεπτά. Παρακαλώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Παρατηρώντας την κατάσταση στην Αλβανία, αισθάνομαι πραγματικά πολύ μεγάλη λύπη, γιατί ανατρέχω στην ιστορία της δικής μου χώρας, τη δεκαετία του 80 κάπου 30 χρόνια πριν, όπου είχαμε πανεφερή κατάσταση. Πάρα πολλέ μεγάλε εντάσει, διαχωρισμού πολιτικές ε, κορυφώσει, απειλέ, ακόμα και βία. Ήταν πραγματικά ένα αποπληκτικό περιβάλλον. Σίγουρα δεν ήμουν υπερήφανο στην εποχή εκείνη. Και κατά τον ίδιο τρόπο, νομίζω ότι οι Αλβανοί πολίτε πρέπει να αισθάνονται ιδιαίτερη λύπη με την όλη κατάσταση στη χώρα του αυτή τη στιγμή. Και εκείνοι σίγουρα δεν είναι περήφανοι για τα τεκτενόμενα αυτή τη στιγμή. Σήμερα είμαι πάρα πολύ περήφανο για τη χώρα μου, γιατί καταφέραμε να δημιουργήσουμε μια χώρα που είναι σταθερή, δημοκρατική και, και πάνω και πρωτίστω από οτιδήποτε άλλο είναι μέλος ευρωπαϊκής οικογένειας. Το πολιτικό περιβάλλον έχει αλλάξει άρδιν. Η δική μου επιθυμία σήμερα είναι ότι και η Αλβανία θα φτάσει θα επιτύχει το στόχο της, γίνει σταθερή χώρα και να είναι μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας. Προφανώς όμως, μέχρι ότου τα δύο κορυφαία πολιτικά κόμματα εξακολουθήσουν να δείχνουν αυτή την ε, απροθυμία και αυτή τη χειρογνωμοσύνη, η Αλβανία θα απέχει πολύ από το στόχο αυτό. Η Ευρώπη κάνει ό,τι είναι δυνατόν μόλις είραμε την απέτηση για βίζα για τους ε, Αλβανούς πολίτες. Αλλά και η Αλβανία πρέπει να κάνει και να αναλάβει τη δική της ευθύνη. Και γι' αυτό πρέπει τόσο η κυβέρνηση όσο και η μείζων αντιπολίτευση να υιοθετήσουν τελείως διαφορετικές πολιτικές, τελείως διαφορετική προσέγγιση που θα είναι όριμες και υπεύθυνες απέναντι στον, Ευρωπαϊκό, στον λαό θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη ενότητα στη χώρα. Δεν είμαστε εδώ βέβαια για να παγορεύσουν του Αλβανού τι πρέπει να κάνουν. Είμαστε εδώ για να του πούμε ότι η απόφαση πρέπει να οδηγήσει την Αλβανία στην ευρωπαϊκή οικογένεια, γιατί εδώ ανήκουν. Ευχαριστούμε πολύ. Περνάμε στην ε, διαδικασία Catch the Eye. Στην αρχή, για ένα λεπτό, η Βρεσάκητς κύριε Πρόεδρε. Eh, Αν και η κρίση στην Αλβανία διαρκεί εδώ και αρκετό διάστημα, τώρα βλέπουμε τις πρώτες μεγάλες κλιμακώσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη φορά ευτυχώς αντέδρασε άμεσα και σωστά κύριοι Φιούλη και Λάιτσεκ αμέσω ανέλαβαν το θέμα και αυτό αποδεικνύει ότι η Αλβανία δεν είναι μόνη τη στην προβληματική αυτή κατάσταση γιατί πραγματικά είναι ένα πρόβλημα που ε, πλήττει την αξιοπιστία της χώρας, ε, μιας χώρας η οποία προσεγγίζει με αξιό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το θέμα δεν είναι εδώ πέρα να δούμε ποιος έχει δίκιο και ποιος άδικο. Πρέπει να δούμε πώς θα επανακαταθέδρυθεί ένας ε, ρεαλιστικός πολιτικός διάλογος και στα πλαίσια αυτά δεν θα έπρεπε να, να ψάχνουμε ποιος έχει δίκιο και ποιος άδικο. Οι δημοτικές εκλογές του Μαΐου θα πρέπει να στείλουν πραγματικό σήμα. Ένα δρόμο προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ή αντίθετο προς την απομόνωση. Ευχαριστούμε πολύ. Είσαι για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, θα συμφωνήσω η σεπήρωση των ανησυχιών των συναδέλφων προηγουμένω, όντω η κατάσταση στην Αλβανία είναι ανησυχητική και θα μπορούσε να έχει αρνητικό αντίκτυπο στι μελλοντικέ προοπτικέ όχι μόνο τη Αλβανία αλλά και όλων των όμορων χωρών. Πέρσι η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέφρασε την άποψη ότι η Αλβανία και η Βοσνία Ζεγοβίνη ε, σημείωναν πρόοδο στη διαδικασία μεταρρύθμισης και απελευθέρωσαν το καθεστώς της Βίζα. Αλλά λίγου μήνε μετά ξεκίνησε πολιτική αναταραχή και υπήρχαν και ανθρώπινες απώλειες. Γι' αυτό ίσως ε, πρέπει να δούμε και πρέπει να ξανασκεφτούμε περαιτέρω τις περαιτέρω προοπτικές περιοχές, γιατί μάλλον η Αλβανία δεν πέρασε το τεστ. Γι' αυτό και όλες οι χώρες στη Βαλκανική περιοχή πρέπει να λειτουργήσουν με έναν αλληλέγυωστό τρόπο και να ενθαρρυνθεί η ένταξη της περιοχής και να στηριχθεί η σταθερότητα. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Η κατάσταση στην Αλβανία, η οποία πραγματικά ήταν εξαιρετικά δύσκολη στην τον Ιανουάριο αποδεικνύει πόσα βήματα έχει ακόμα να κάνει η χώρα. Ξέρετε ότι είχαμε, θρυνήσαμε θύματα και νομίζω ότι σε δημοκρατικά καθεστώτα τέτοιου είδους αντιδράσεις δεν θα πρέπει να οδηγούν σε ταραχές ε, και σε επεισόδια, αλλά θα πρέπει να λύνονται ελεκτικά στο Κοινοβούλιο. Το γεγονός ότι κάποιες από τις αρχές ε, προσπαθώντας να καλύψουν τους ενόχους ε, συμπεριφέρθηκαν με τόσο αξιοθρύνητο τρόπο, νομίζω ότι θα πρέπει να καταδικαστεί. Οι εκλογές του 2009 ε, θα πρέπει να γίνουν σεβαστές γιατί όλοι συμφώνησαν πως τότε οι εκλογές έγιναν με άμετο τρόπο. Οπότε νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να το τονίσουμε. Ευχαριστούμε πολύ κ. Πανικολάου για ένα λεπτό. Ήθελα να κάνω την εξής επισήμανση. Προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι ενώ οι δείκτες ανάπτυξης στην αλβανία είναι σταθερά ανωδικοί και θυμίζω ότι εν μέσω παγκόσμιας οικονομικής αστάθειας η ανάπτυξη στη χώρα ξεπέρασε το 2% το 2010 και για το 2011 η πρόβλεψη είναι να φτάσει το 3% παρόλα αυτά οι κοινωνικές εντάσεις οξύνονται αντί να αμβλύνονται. Και είναι προφανές, κύριε Επίτροπε, ότι η ανάπτυξη δεν έχει εμφυτεύσει στους Αλβανούς πολίτες το αίσθημα της ευημερίας αντίθετα είναι προφανές επίσης ότι αυξάνεται η απογοήτευση και μαζί της και η φόβοι για ένα νέο κύμα μετανάστευσης των πολιτών της προς γειτονικές χώρες αφού το ζήσαμε πολύ έντονα τη δεκαετία του 90 στην ελλάδα. σε τούτη λοιπόν τη δύσκολη στιγμή χρέος της ευρώπης είναι εκτός από τις πολιτικές παρενέσεις προς την αλβανία να στηρίξει εμπράκτος, να μεταφέρουμε πρακτικές και παραδείγματα ώστε η ανάπτυξη να αποβεί προς όφελος όλων των κοινωνικών ομάδων. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τέλος, τελευταίος αλλογή. Ελλάσσον ο κύριος Σουέφιλ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα συνεχίσω στα αγγλικά. Η κατάσταση αυτή περιγράφεται ως ψυχρός εμφύλιος. Τα πολιτικά κόμματα είναι οι εμπόλεμοι και οδηγούν τη χώρα σε μια αρνητική δίνη. Η εξήγηση είναι πως αριστερά και δεξιά πιστεύουν πως τα πολιτικά κόμματα θα πρέπει να κυβερνούν αποκλειστικά όπως έκανε κάποτε το Κομμουνιστικό Κόμμα. Μόλις έχει ξεκινήσει λοιπόν αυτή η πόλωση είναι πάρα πολύ δύσκολο να αλλάξει η κατάσταση και να γίνει μια κατάσταση που μοιάζει με δημοκρατία γιατί βεβαίως η αποκλειστική εξουσία όπως το βλέπουν στην Αλβανία είναι κάτι το απολύτως λογικό και αυτό είναι τραγικό. Υπάρχει διέξοδος, ναι, κάθαρση αλλά μόνο μια μεγάλη κρίση, ένας μεγάλος ιστορικός συμβασμός μπορεί να προκαλέσει κάτι τέτοιο. πολύ. Και για το ότι τηρήσατε και το χρόνο σας πέραν όλων των άλλων. Ήταν ο τελευταίος ομιλητής στον κατάλογο μου και τώρα ζητώ από τον Επιτροπή Φίλε να συνοψίσει όλα όσα συζητήθηκαν αυτή τη στιγμή. Thank you very much. Uh, Mr. President, honorable members. Uh, Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, να σας ευχαριστήσω για αυτή τη συζήτηση, την έντονη συζήτηση. Και πριν περάσουμε στις παρατηρήσεις μου, θα ήθελα να αναφερθώ στα δύο ερωτήματα που μετέθησαν. Το πρώτο, τον κύριο Μπέλντνερ, θα το απαντήσω γραπτός λαμβάνοντας υπόψη το ότι σήμερα εστιαζόμαστε αλλού. Α, υπήρχε κι άλλο ένα ερώτημα. Το εάν σκεφτόμαστε κυρώσεις. Όχι. Δεν σκεφτόμαστε κάτι τέτοιο. Γιατί, γιατί στην διεύρυνση οι προϋποθέσεις λειτουργούν σαφώς και δίκαια. Αν όταν εκπληρώνει κανείς προϋποθέσεις, προχωρά μέχρι να ενταχθεί στην Ένωση. Αν δεν εκπληρώνει κανείς τις ε, προϋποθέσεις, επιβραδύνει και σταματάει. Δυστυχώ, αυτό είναι το τίμημα που πληρώνουν τώρα όχι μόνο οι πολιτικοί, αλλά και οι πολίτες της χώρας αυτής. Κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, η είπατε εκπρόσωπος και εγώ θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες για να συνεχιστεί ο διάλογος μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης στην Αλβανία. Έχουμε μια σαφή ιδέα για το πώς θα γίνει αυτό. Χρειαζόμαστε και τη δική σας στήριξη για να διασφαλίσουμε πως ε, ο ηγέτης αντιπολίτευσης και ο πρωθυπουργός της χώρας ε, να αντιληφθούν το μήνυμά μας. Έτσι μπορεί να φύγει η χώρα από την πολιτική κρίση και να γίνουν θετικά βήματα προς την ευρωπαϊκή της ένταξη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναλάβει μια δέσμευση εναντί όλων των χωρών των Δυτικών Βαρκανίων πώς να ενταχθούν στην Ένωση. Τηρούμε αυτή τη δέσμευσή μας και θα αυξήσουμε την εμπλοκή μας αρκεί να εκπληρώσουν τα κριτήρια οι χώρες. Η Αλβανία χρειάζεται επιγόντω να εφαρμόσει τις 12 προτεραιότητες κλειδιά της Ένωσης. Αυτές συμπεριλαμβάνουν τις θεμελιώδεις αρχές της δημοκρατίας, όπως η σωστή λειτουργία του Κοινοβουλίου, ο διαχωρισμός των εξουσιών, εξαγωγή εκλογών και σεβασμός του κράτους δικαίου. Όλα αυτά θα είναι δυνατά μόνο όταν ε, μεταβληθεί προς το καλύτερο η πολιτική κατάσταση με την επανάληψη πολιτικού διαλόγου στο Κοινοβουλίο Σεβασμού των θεσμών του κράτους και όταν συνειδητοποιήσουν πως οι πολίτες της Αλβανίας έχουν φιλοδοξίες που χρειάζονται την προσοχή τους και οι ηγέτες της Αλβανίας πρέπει να δράσουν τώρα για το καλό του λαού τους και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να τους βοηθήσει. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, ελπίζουμε η κατάσταση στην Αλβανία να εξομαλυνθεί και κλείνω τη συζήτηση με αυτή την ιδέα και συνεχίζουμε με το επόμενο θέμα της σημερινής διάταξης που είναι η δήλωση της Επιτροπής αναφορικά με το σκάνδαλο υποκλοπής κλήσεων στη Βουλγαρία.